την ολοκληρώσαμε έτσι και η ψηφοφορία θα λάβει στις Βρυξέλλες χώρα. Κυρίε και κύριοι, προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης σε μια προφορική ερώτηση συγκεκριμένα για προφορική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα της ασφάλειας των αερομεταφορών, μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εναέρειες μεταφορές. Και το λόγο λαμβάνει πρώτη η κυρία Τσικάου, η συντάκτρια της προφορικής ερώτησης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα περιμένω μερικά δευτερόλεπτα. Thank you, Madam Chair. Mr. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Πίλμπαρξ. Η ερώτηση υπευλήθη από τον Brian Simpson εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών του Τουρισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής ε, για το θέμα της μαύρης λίστας. Η μαύρη λίστη, λίστα ε, συστάθηκε το 2005 και αφορούσε τις ε, επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις διεθνείς κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα. Μετά από κάποιες κάποια δυστυχήματα το 2004-2005. Εδώ τέσσερα χρόνια ξέρουμε ότι η μαύρη λίστα έχει αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την επιβολή των κανόνων ε, στι διεθνεί οργάνωση τη πολιτική αεροπορία, προστατεύοντα και τους Ευρωπαίου πολίτε. Αυτό το οποίο μα προβληματίζει σήμερα είναι το εξή. Πώ θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε αυτήν την ασφάλεια και να εργαστούμε περαιτέρω για την βελτίωση των κανόνων ασφαλείας. Η μαύρη λίστα δεν αφορά μόνο το που βρίσκονται οι κίνδυνοι για τους επιβάτες, αλλά να διασφαλίσει ότι και οι πληροφορίες φτάνουν στα χέρια των Ευρωπαίων πολιτών. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίες παίρνουν πτήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, θα επιβιβαστούν σε αυτές τις εταιρείε που συνεχίζουν να εκτελούν τόσο εσωτερικέ πτήσει όσο και άλλε πτήσει σε περιοχές του κόσμου και έτσι βρίσκονται στη μαύρη λίστα. Πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι οι επιβάτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργηθεί μία ενιαία και μοναδική μαύρη λίστα, αλλά η μαύρη λίστα φυσικά είναι και η μοναδική δυνατότητα που έχουμε προκειμένου να ε, ενημερώσουμε τους πολίτες μας. Πώς μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε σε αυτούς, αυτή τη μαύρη λίστα και να είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις ε, πληροφορίες αυτές και ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να δυσπρίσει ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις στον τομέα της ασφάλειας βάσει των ελέγχων της ε, Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής αεροπορία. Ε, τώρα, επί φορά φορές προφορίες που βρώνουν από τρίτε χώρε, η Κομισιόν προτίθεται να ε, υλοποιήσει ένα σύστημα για ανταλλαγή αξιόπιστων στοιχείων που θα ε, στηρίζονται στις ε, διάφορες μαύρες λίστες ε, που υπάρχουν. Επίσης θα θέλαμε να πούμε ότι η μαύρη λίστα έχει αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο προκειμένου να υποχρεώσουμε κάποιες αεροπορικές εταιρείες να τηρήσουν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Και πώς η Κομισιόν λοιπόν προτίθεται να υποστηρίξει τις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας προκειμένου να καλύψουν τα κενά που έχουν σε θέματα ασφάλειας και να συμμορφωθούν απόλυτα με το Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. Χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τους πολίτες, αλλά και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να, να εργαστούμε ώστε ε, να βελτιώσουμε περαιτέρω τα πρότυπα ασφάλειας. Αυτό θα ήταν ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να υπάρξει ασφάλεια για όλους τους πολίτες. Η Επιτροπή ε, Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου επιθυμεί να συνεργαστεί με την Κομισιόν προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξενόματος της Επιτροπής. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Πίμπαλξ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τσίκαου για την ε, θετική της προσέγγιση για τις μαύρες λίστες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι ε, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενημερώνουν πάρα πολύ σωστά το κοινό για τις πτήσεις από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κατάλογος των αεροπορικών εταιριών που απαγορεύεται να κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και ε, στο διαδίκτυο αλλά και με στοχευμένες δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με την ΙΑΤΑ κάθε φορά ε, που ανημερώνει το κατάλογος αυτός για να έχουμε την καλύτερη δυνατότητα ενημέρωσης των επιβατών. Οι ε, αρχές πολιτικής αεροπορίας και ε, των αερολιμένων των κρατών μελών είναι υποχρεωμένες να θέτουν στη διάθεση των πολιτών και των επιβατών ε, αυτές τις προφορίες και στην ιστοσελίδα τους αλλά και επί τόπου Η λίστα ε, δίνει χρήσιμες προφορίες στους επιβάτες που θα ταξιδεύουν και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφεύγουν να τις χρησιμοποιούν. Δεν έχει βέβαια κανένα χαρακτήρα ετεροδικίας ούτε μπορεί να βρει εφαρμογή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η λίστα αυτή. Αλλά καλό είναι ε, να λέμε ότι οι ε, επιβάτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν με ποια εταιρεία ε, ταξιδεύουν και κάθε ταξιδιωτικός πράκτορας ή tour operator είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τη στιγμή της κράτησης στον επιβάτη ποιες εταιρείες ενέχονται στην πτήση αυτή. Και ε, ε, επίσης σε περίπτωση αλλαγής εταιρεία θα πρέπει να το γνωρίζει ο επιβάτης. Είτε ε, στο check-in είτε το αργότερο τη στιγμή της επιβίβασής του στο αεροπλάνο. Και να έχει το δικαίωμα αποζημίωσης ή αλλαγής δρομολογίου αν έχει αλλάξει η εταιρεία σε περίπτωση που ακυρωθεί η πτήση του. Επίσης υπάρχουν και διάφορες πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε αν συμμορφώνονται στις διεθνείς διατάξεις οι εταιρείε. Έλεγχοι ασφαλείας γίνονται από τον ΑΙΚΑΟ. Επίσης ε, δίνονται προφορίες από τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών καθώς επίσης και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Πολιτικής ε, Αεροπορίας στα πλαίσια των ελέγχων και των επιθεωρήσεων που κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και σε τεχνικές αποστολές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται επίσης τυχαίοι έλεγχοι ε, ε, στα πλαίσια αντίστοιχου προγράμματος αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σύμφωνα με τους κανόνες και επίσης ε, δίνεται στοιχειοθετημένη, τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε σχέση με τα αεροπορικά δυστυχήματα ω απόρρια των δυστυχημάτων αυτών. Επίση, θα πρέπει να σα πω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εξαντλητικό κατάλογο χωρών που έχουν αντίστοιχη νομοθεσία, αλλά υπάρχουν ε, ε, ε χώρε όπω ε, το Μπαχρέιν, η Δημοκρατία τη Κορέα ή το Βασίλειο τη Σαουδική Αραβία έχουν αντίστοιχου κανόνε με την Ευρωπαϊκή Λίστα. Επιβεβαιώνω και πάλι την προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο για τη νομοθεσία αυτό, για να υπάρχει ε, μεγαλύτερη ασφάλεια των πτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Πρώτη κυρία Ντεβεράκ, παρακαλώ, για δύο λεπτά. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπήρξα εισηγήτρια πριν από πέντε χρόνια για αυτόν τον κανονισμό και χαίρομαι που διαπιστώνω ότι ε, εφαρμόζουμε ένα μηχανισμό ο οποίος λειτουργεί και έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Η έκθεση της Κομισιόν για την εφαρμογή του κανονισμού για τον Μαύρη Λίστα νομίζω ότι είναι πλήρη. Προτείνει κάποιες, ε, ενδιαφέροντε προ, προβληματισμούς, εγώ συμφωνώ ότι μια παγκόσμια μαύρη λίστα θα είναι μοναδική εγγύηση για την ασφάλεια των αεροσκαφών. Θα ήθελα να θέσω όμως κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Θα ήθελα να μάθω πώς γίνεται ο έλεγχος των ε, διαφόρων ε, εταιριών ε, ελέγχονται, δηλαδή γίνεται ακρόαση με τις, αρχές, με τις εταιρείες αυτές ή μόνο με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το εξασφαλίσουμε. Επίσης κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό είναι το θέμα της παρακολούθησης των αεροσκαφών. Η Κομισιόν παρακολουθεί τα αεροσκάφη μιας αεροπορικής εταιρεία που έχουν μπει στον μαύρο πίνακα ή από τον οποίο έχουν αποσυρθεί κάποια πιστοποιητικά προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα αεροσκάφη αυτά δεν πετούν με άλλο όνομα, με άλλες εταιρείε και να μην υπάρχουν ε, ένα είδος σημαίων ευκαιρίας λοιπόν και στην περίπτωση της ε, αεροπλοείας. Στην περίπτωση λοιπόν που μια εταιρεία μπαίνει στο Πίνακα, η Κομισιόν λαμβάνει πληροφορίε αναφορικά με τον ποιο τρόπο ενημερώνουν οι πράκτορες ε, ταξιδίων τους πελάτες τους και τι εναλλακτικές λύσεις προτείνουν και καμία συγκεκριμένη περίπτωση. Πολλοί βουλευτές λάβαμε μηνύματα σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Ινδονησίας όπου όλες οι εταιρείες έχουν απαγορευτεί και μας ζητούν να παρεύουμε προς την, και να επηρεάσουμε την Επιτροπή έτσι ώστε να αρθούν αυτοί οι αυτές οι απαγορεύσεις. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς έχει κατάσταση στην χώρα αυτή τώρα διότι εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται στο μαύρο πίνακα και αν η Ινδονησία έχει καταβάλει προσπάθειες για να μειώσει, να καταργήσει τις ελλείψεις θέματα ασφάλειας. Ευχαριστώ κύριο Σαχαντράουι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Για δύο μισή λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι λίγο σουρεαλιστικό να συζητάμε τώρα τέτοια πράγματα για τη μαύρη λίστα τη στιγμή που πολλές αεροπορικές εταιρείες και η αεροπορία γενικά στην Ευρώπη έχει παραλύσει και είναι χάος. Αλλά από ό,τι κατάλαβα αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε επίκαιρη συζήτηση και θα λάβω και το λόγο. Η μαύρη λίστα αυτή καθ' αυτή είναι σημαντικό ζήτημα και μπορούμε να πούμε και επιτυχία πλέον μεταξύ άλλων χάρη στην όθηση της κυρίας Δεβεράκ που πριν από λίγα χρόνια άρχισε να δουλεύει και δούλεψε πολύ σκληρά. Λέω επιτυχία γιατί ε, εξάγουμε διδάγματα από την εμπειρία του παρελθόντος. Και βεβαίως χρειάζονται και νέες προσπάθειες και από πλευράς ενημέρωσης προς τους επιβάτες. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να ενημερώνονται οι επιβάτες και από τα ταξιδιωτικά γραφεία και τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί το ποιες εταιρείες είναι στη Μαύρη Λίστα, αλλά συχνά οι επιβάτες αποφασίζουν μόνο ε, επιτόπου ε, ή μπορούν να αποφασίσουν για μια πτήση εσωτερική αν ε, θα πάρουν την πτήση αυτή ή όχι. Και θα ήθελα να πω το εξής. Κάποια πρακτορία που κλείνουν ταξίδια για χώρες που λειτουργούν τέτοιε επισφαλείς εταιρείε θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τους επιβάτες πριν ξεκινήσουν ότι εκεί λειτουργούν τέτοιες εταιρείες. Και ένα δεύτερο στοιχείο θα πρέπει να συμβάλλουμε στην αποφυγή ε, συμπερίληψης ε, και άλλων εταιριών και άλλων χωρών στη λίστα αυτή. Θα πρέπει να βοηθούμε τις φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους υποστηρίζουμε έτσι ώστε και οι δικές τους αεροπορικές αρχές, αρχές ενέργειας κυκλοφορίας να έχουν ε, τη δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Βέβαια, είπε η κυρία Ντεβεράκ ότι υπάρχει και κάποιο πρόβλημα παραπληροφόρησης. Αν υπάρχουν δυνατότητες παραθυράκια να ξεφύγει κανείς από, ε, που είναι στη μαύρη λίστα, ε, να λειτουργεί σε άλλη χώρα με άλλο όνομα, τα ξέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και ένα τελευταίο, θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια παγκόσμια μαύρη λίστα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι προσπάθειες έχετε κάνει προς την κατεύθυνση αυτή του ΑΙΚΑΟ, ας πούμε, με τους συναδέλφους ομολόγους σας από άλλες χώρες, για να υπάρχει παγκόσμια πλέον λίστα. Ευχαριστώ. Μάισνερ από τους φιλελευθέρους για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι τώρα έχουν μείνει ακινητοποιημένα όλα τα αεροπλάνα, ότι δεν υπάρχουν πτήσει στου ευρωπαϊκού ουρανού. Είναι ένα θέμα το οποίο μα έχει απασχολήσει. Είναι ταυτόχρονα κάτι το οποίο έχει και οικονομικέ επιπτώσει και θα πρέπει να το δούμε μέσα από την οικονομική αυτή διάσταση. Ταυτόχρονα όμω διαφυλάσσοντα και την ασφάλεια, γιατί έχουμε να κάνουμε την ασφάλεια των αερίων μεταφορών των Ευρωπαίων ε, επιβατών. Είναι πολύ σημαντικό για μας στην Ευρώπη να μπορεί ο καθένας να αποφασίσει ελεύθερα το πώς θέλει να μετακινηθεί, με ποια αεροπορική εταιρεία θέλει να κάνει την κράτησή του και με ποια δεν θέλει. Και για να μπορέσει να αποφασίσει κανείς ελεύθερα πρέπει να έχει επαρκείς πληροφορίες στη διάθεσή του και στην ουσία. Μαθαίνουμε λοιπόν το 2006 Ήδη καταρτίστηκαν αυτές ε, οι μαύρες λίστες και θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί για το αν ε, μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν τα αεροπλάνα αυτά ή όχι. Αλλά το κύριο ερώτημα για μένα είναι και αυτό του τη κυρία Ντεβεγά και του κυρίου Λιχαντράου. το αν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι πως δίνονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητε για την ασφάλειά μα βεβαίω καταρχά. Θέλουμε όλοι οι επιβάτε εδώ στην Ευρώπη να έχουν ασφαλείς συνθήκε πτήσεω. και δεύτερον, ιδιαίτερη σημασία θα έχει πιστεύω, και το να γνωρίζουμε με ασφάλεια το αν είναι και αρκετά στεναρή οικονομική, οικονομικά μία ε, αεροπορική εταιρεία. Γιατί πολλές φορές επιτρέπεται η λειτουργία αεροπορικών εταιριών ε, όχι μόνο για λόγους ασφάλειας, ε, δηλαδή ε, γιατί έχει ασφαλή αεροπλάνα και μπορεί να διεξαγάγει ασφαλείς πτήσεις, αλλά θα πρέπει να ελέγχει ταυτόχρονα και η οικονομική ασφάλεια, δηλαδή το ότι θα μπορεί να συνεχίσει να πετά ε, τα αεροπλάνα τη και ότι δεν θα κηρύξει πτώχευση ανα πάσα στιγμή. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είδαμε πέρσι με τη Sky Europe, με Ευρωπαίου πολιτέ οι οποίοι είχαν κάνει τι κρατήσει του αεροπλάνα. Δεν είχαν καμία ενημέρωση ότι βρισκόταν αυτή η εταιρεία στα πρόθυρα τη πτώχευση και όταν ήρθε η στιγμή βρέθηκαν ε, αποκλεισμένοι σε αεροδρόμια χωρί καμιά ενημέρωση και πάνω απ' όλα χωρί καμιά προστασία. Και γι' αυτό θα ήθελα να γνωρίζουμε, όταν ε, μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να έχει πληροφορίε, θέλουμε να ξέρουμε ότι μπορεί να διαθέσει τι πληροφορίε αυτέ και στο κοινό γιατί δεν δημοσιεύτηκαν αυτέ οι πληροφορίε και πώ μπορούμε να έχουμε εξασφάλιση ότι πάντοτε θα είναι διαθέσιμες οι απαραίτητε πληροφορίε στον επιβάτη. Και γι' αυτό θα ήθελα να, γίνουν, να δοθούν και σχετικέ απαντήσει στη συζήτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Η επόμενη ομιλήτρια εκ μέρου των Πρασίνων είναι η κυρία Λίχτενμπεργκερ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το Κοινοβούλιο όταν συζητήθηκε η κατάρτιση των μαύρων ληστών, των ε, αρνητικών καταλόγων, είχε καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον Ευρωπαίο επιβάτη. Βέβαια, τώρα το ζήτημα, εάν όπως έχουν τώρα οι συνθήκες, είναι επαρκής αυτή η ε, ασφάλεια, η παρεχόμενη ασφάλεια. Και θα ήθελα να συστήσω το θέμα ως προς το εξής. Ναι, οι πληροφορίες που διαθέτεται μέσω του ίντερνετ είναι διαθέσιμες μεν, αλλά, όχι δεν είναι αλλά δεν είναι και τόσο ευανάγνωστες για τον κοινό ε, επιβάτη, ιδιαίτερα για ορισμένε αεροπορικέ εταιρείε, δεν είναι καθόλου εύκολο να τι βρει κανεί. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πτήσει μέσω μια διαφορετική ε, εταιρεία που αναλαμβάνει μια τρίτη εταιρεία ή που περνούν μέσα από τρίτο κράτο. Πρώτον. Δεύτερον, Πώς, γίνεται η... πώς βλέπετε τα πράγματα σχέση με το wet leasing, ποια είναι οι εμπειρίε που έχουμε από αυτό το σύστημα. Μήπως αυτό τελικά αποτελέσει και το παραθυράκι ώστε να μπουν όχι τόσο αξιόπιστες επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες δηλαδή στους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ήδη από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας. Και Τρίτον, οι διατάξει αυτέ για την μαύρη λίστα δεν θα πρέπει να έχουν και προληπτικό χαρακτήρα για αεροπορικέ εταιρείε οι οποίε δεν έχουν τηρήσει το παρελθόν και έξω και από την Ευρώπη τι ε, ε, προποθέσει ασφαλεία. Πρώτον και δεύτερον, πώς γίνεται επιλεκτικά να επιτρέπεται η ε, κυκλοφορία συγκεκριμένων αεροσκαφών ε, μια εταιρεία, ενώ κάποιες άλλες της ίδιας εταιρείας, ε, κάποια άλλη τη εταιρεία δεν επιτρέπεται να πετούν στου ευρωπαϊκού ουρανού. Ευχαριστώ, κύριο Σαρνέσκι, τώρα από του Ευρωπαίου Στερετικού και Μεταρρυθμιστέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμα μέλη, δεν είμαι διόλου βέβαιος πως ε, οι επιπτώσεις του ηφαιστείου της Ισλανδίας θα πάψουν σύντομα να μας ε, επηρεάζουν και να ταλαιπωρούν τους ε, πιβάτες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό το γεγονός και στις ε, τιμές τις οποίες θα κληθούν να πληρώσουν οι επιβάτες ε, των αεροπορικών μεταφορών. Το ζήτημα λοιπόν αυτό που μας απασχολεί τώρα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Επαντηλημένα έχω μιλήσει για το ζήτημα αυτό στο ε, σημερινό κοινοβούλιο αλλά και στο προηγούμενο. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Ένας Πολωνός δημοσιογράφος πρόσφατα με ρώτησε τι κάνετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτές τις ε, περιπτώσεις. Το ζήτημα της ασφάλειας είναι ζωτική σημασίας. Και αυτό είναι προς όφελος ε, των πολιτών μας, των καταναλωτών μας ε, και όλων των υπολείπων. Γι' αυτό και τα μέσα ενημέρωσης ενδιαφέρονται το κατά πόσον το θέμα αυτό μας αποσχολεί. Γνωρίζουμε πως υπάρχει αυτή η μαύρη λίστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι σαφές το ποιες αεροπορικές εταιρείε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται σε αυτή τη μαύρη λίστα. Δεν θα πρέπει οι πολίτες να πληρώνουν επιπλέον για την ασφάλεια Τώρα οι λοιποί ομιλητές, ο κύριος Γκρός, πρώτος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η μαύρη λίστα ήταν ενδιαφέρον επίταγμα ε, του Κοινοβουλίου υπό την ηγεσία της και Κριστίν Ντεβεράκ και τους άλλους συναδέλφους στην προηγούμενη θητεία. Αυτό μπορεί να αφορά εταιρείε, κράτη ή αεροσκάφη η λίστα. Γι' αυτό θα ήθελα να μας απαντήσει πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χώρες. Ποιο είναι το δικαίωμα λόγου που έχουν οι συναπόφαση οι εταιρείε. και όταν πρόκειται για μεμονωμένα αεροσκάφη, για ποιο λόγο γίνεται αυτό και πώς έχει η διαδικασία. Ήδη πριν από λίγα χρόνια τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά και εξηγήσαμε και παραμένει για μας σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο θέμα αυτό και να παρακολουθήσει και ε, το νομοθέτημα και τα μέτρα και στην επικοινωνία με το Κοινοβούλιο να βελτιωθεί η, ε, η πληροφόρηση γιατί για, για μας παραμένουν ορισμένα ζητήματα ε, σε κρεμότητα. Πώς μπορούν να αλλάξουν όνομα οι εταιρείε ή για τα αεροσκάφη ακόμα για να εξακολουθούν να ε, πετάνε και αποφάσεις τελευταία στιγμής. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, απαιτούν τη στοιχειώδη διαφάνεια. Και ένα σημαντικό για μένα θέμα είναι η ενημέρωση, η πληροφόρηση. Εμείς θεωρούμε γενικά, νομίζω σε όλες τις πολιτικές ομάδες, ότι οι πολίτες και οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα, άρα και υποχρέωση ε, των εταιριών να τους ενημερώνουν συστηματικά για τις μαύρες λίστες και ε, να ε, μπορεί κάθε επιβάτης να την προμηθεύεται στα αεροδρόμια και στα ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συγκεκριμένε χώρες εντός εισαγωγικών που είναι ήδη γνωστές ως προβληματικές, να ε, το εξηγούν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ποιες είναι οι εταιρείε προβληματικές σε περίπτωση που χρειαστεί κανείς να αλλάξει το εισιτήριό του. Μπορεί να έχει βελτιωθεί η ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί ε, ο κατάλογος αυτός και να καλύψει τον κόσμο όλο, όχι μόνο την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους επιβάτες. Ευχαριστώ. Η Φιώνα Χόλ για δύο λεπτά παρακαλώ, επόμενη μιλήτρια. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλεια των αέριων μεταφορών και που υπογραμμίζει την ανάγκη η, ο, ο, η μαύρη αυτή λίστα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί λειτουργική το χέτερο δυνατό. Το 2008 το, το Συμβούλιο εν τέλει υιοθέτησε τον κώδικα συμπεριφοράς Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταφορά όπλων που ελέγχει την εξαγωγή τέτοιου είδους ε, πολεμικού υλικού. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλέ ανησυχίε ότι δεν τηρούν αυτόν τον κώδικα συμπεριφοράς όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που εξαγούν όπλα, εξαγωγή όπλων. Ένα μέτρο απεδείχθη ιδιαίτερα σημαντικό δε για τον, ε, για τον έλεγχο της ε, λαθρέας ε, πόλης όπλων και αυτό ήταν η μαύρη λίστα. Με μια μελέτη που έγινε το 2008 αποδείχθηκε ότι ενέργειες μεταφορές, οι οποίοι ήταν ε, μεταφορές που ήταν εμπλεγμένοι σε εμπόλεμες ζώνες, ήταν ταυτόχρονα και εκείνοι οι οποίοι επανελειμμένως παρεβίαζαν τις συνθήκες ασφαλείας. Ίσως είναι και λογικό εκείνοι οι οποίοι δεν υπολογίζουν ιδιαίτερα τις συνθήκες ασφαλείας να μην ενδιαφέρονται και ιδιαίτερα για το τι φορτίο μεταφέρουν. Πάντως η συνέπεια αυτής της συνδυασμένης παρέμβασης σημαίνει ότι μέτρα τα οποία έχουν σαν πρόθεση ή σαν στόχο να προστατεύσουν τον Ευρωπαίο πολίτη εξυπηρετούν ταυτόχρονα και την προστασία και άλλων πολιτών, της Αφρικής ιδιαίτερως, από, τα καταστροφικά, από τις καταστροφικές συνέπειες των όπλων, ελαφρών όπλων, ελαφρού οπλισμού που συχνά πωλείται από ευρωπαϊκά κράτη κατά τρόπο παράνομο. Παρακαλώ λοιπόν και τον κύριο Επίτροπο να πιέσει ο ίδιος και να βοηθήσει στις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τακτική και συστηματική τήρηση των μαύρων αυτών ληστών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζιόμπρο πάλι δεν είναι εδώ παρόν. Ο κύριος Μαρινέσκου έχει το λόγο δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή η μαύρη λίστα των αερομεταφορέων είναι πράγματι ένα πολύ θετικό μέτρο για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να ε, διευρυνθεί και να ε, δημοσιεύεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο αλλά και από τα ταξιδιωτικά γραφεία, από τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Ταυτόχρονα χρειάζεται να βρεθούν και λύσει σε περιπτώσει όπου υπάρχει μία και μόνο αεροπορική σύνδεση με μία μόνο εταιρεία, η οποία όμω έχει μπει στη μαύρη λίστα. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδου λίστε. Πολλέ από τι επιχειρήσει τη μαύρη λίστα ξέρουμε ότι πετούν σε υποανάπτυκτα τρίτα κράτη της ε, Αφρικής ή της Κεντρικής ή Ασίας και γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα πώς μπορεί να εξασφαλιστεί και ο ε, θεμητός ανταγωνισμός, ο επίσης ο ανταγωνισμός μεταξύ των αεροπορικών εταιριών ε, αυτών και εκείνων της Ευρώπης, ε, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και των άλλων σοβαρών ε, αεροπορικών εταιριών. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε και μια ε, δίκαιη κατανομή των σχετικών αδειών ανά τον κόσμο. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει και στην ανάπτυξη όλων των κρατών. Καλώ λέει η πρόεδρο, ευχαριστώ. Περνούμε στη δικασία του Καρστία Διάη. Ο κύριο Λάιχτφριντ έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ε, μια γενική παρατήρηση έχω και δυο τρει ερωτήσει ανάλογα με το χρόνο που θα μου ε, δώσετε. Η γενική παρατήρηση. Μου φαίνεται λίγο μυστήριο περίπου το γεγονός ότι στη σημερινή κατάσταση ως σοσιαλδημοκρατική ομάδα σε τρεις εκθέσεις για την ασφάλεια στις αερόμεταφορές έχουμε συνολικά 9 λεπτά χρόνο. Το καταλαβαίνω ότι είναι έκτακτες οι περιστάσεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε χρόνο για να συζητάμε θέματα που ε, ασχολούνται ε, με την καθημερινότητα και τα προβλήματα των πολιτών και σε κάποιες άλλες συζητήσεις να αφαιρώνουμε λιγότερο χρόνο. Θέλω να ρωτήσω κύριε Επίτροπε, τι γίνεται με τις ε, πτήσεις code shared, δηλαδή έχεις ένα με μια εταιρεία και τελικά την πτήση την κάνει μια εταιρεία που μπορεί να είναι και σε μαύρη λίστα. Αυτό είναι πάρα πολύ καυτό ερώτημα που απασχολεί τους πολίτες και θα περίμενα να μου απαντήσετε. Ορίστε, μία ερώτηση έκανα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όμπερ Μάιερ και εκείνο για ένα λεπτά. Αφού μιλάμε για την ασφάλεια στις πτήσεις και μεθαύριο ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Πτήσεων θα θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ε, ρωτήσω κάτι άλλο προβληματικό. Στην Αυστρία, εκεί που κάνουν αέρια ε, αθλήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα υπαρξιακά. Ε, και μας λένε οι αθλητές ε, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ, παρά που μιλούν εξαιρετικά αγγλικά, είναι πολύ δύσκολη η ορολογία ειδική για εκείνους σε άλλες γλώσσες και προσπαθούν να τους ε, βάλουν ε, άχρηστα εμπόδια. Γι' αυτό παρακαλώ ε, οι κανονισμοί που είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τους αθλητές αυτούς να μεταφράζονται και στα γαλλικά και στα γερμανικά στις άλλες δύο γλώσσες εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επόμενη και τελευταία ομιλήτρια στη δικασία του Καρστία είναι πάλι η κυρία Τσίκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η μαύρη λίστα που ε, ενημερώθηκε στις 30 Μαρτίου του 2010 περιλαμβάνει πολλές επιχειρήσεις από 17 κράτη-μέλη και πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει τις δυνατότητες που έχει έτσι ώστε να παρακολουθεί την, ε, τις εξελίξεις ε, και τη συμπεριφορά των αεροπορικών εταιριών, ώστε μόνο αυτές οι οποίες τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές να έχουν το δικαίωμα να πετούν στους ευρωπαϊκούς ε, ουρανούς. Ταυτόχρονα θα πρέπει να βοηθήσουμε και τα τρίτα κράτη, ώστε να βελτιώσουν εκεί οι εταιρείε τις προδιαγραφές τους και τις ικανότητές τους και ταυτόχρονα να τα ενισχύσουμε ώστε να χορηγούν άδεια μόνο, μόνο στις επιχειρήσεις που τηρούν τις σχετικές προδιαγραφές. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάζεται και συγκεκριμένα τι είδους αεροσκάφη ε, χρησιμοποιεί κάποια εταιρεία, αλλά και τι είδους ε, ιστορικό έχει, ε, ιστορικό ατυχημάτων κτλ. Οι υποδομές της επίσης, οι υποδομές της θα πρέπει να ελέγχονται και για την δυνατότητα αγοράς και χρήσης των εισιτήριων. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Πίμπαρεξ, ο Επίτροπος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις σας κυρίες και κύριοι βουλευτές γιατί δείχνουν ότι στηρίζει την προσέγγιση αυτής της μαύρης λίστας στο Κοινοβούλιο και σας διαβεβαιώνω και προσωπικώς και εκ μέρους του Αντιπρόεδρου Κάλλας ότι θα λάβουμε υπόψη όλες τις παρατηρήσεις αποφάσεις που θα λάβουμε και θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ε, απαντώντας βέβαια στις ερωτήσεις, επειδή ήταν πολύ άριθμες, είμαι υποχρεωμένο να επιλέξω μόνο κάποιε από αυτές, διαφορετικά θα μπορούσα να τηρήσω το χρόνο του 1,5 λεπτού. Καταρχά για τα ε, διεθνή, διεθνή διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξετάζει αυτό το θέμα προσπαθώντας με κάθε, ε, με κάθε ευκαιρία να ενισχύει τη διεθνή συνεργασία ώστε κάθε κράτος να ε, κάθε τρίτο κράτος να εντάσσεται στα προγράμματα για την ασφαλή αξιολόγηση και ταυτόχρονα προσφέρει και προγράμματα τεχνικής συνδρομής ε, ώστε κάθε κράτος να αναπτύξει τις απαραίτητες προδιαγραφές, διεθνείς προδιαγραφές. Συνεργαζόμαστε επίσης με την ΙΚΑΟ μέσα δε και από την διάσκεψη που είχαμε το Μάρτιο για τις διεθνείς, για τις διεθνείς ασφαλείς πτήσεις ε, και την περαιτέρω συνεργασία και το πρωτόκολλο που έχουμε υπεγράψει θα συνεχίσουμε βεβαίως αλλά δεν θα πρέπει και να υποτιμούμε την, ε, ε, τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτή η μαύρη λίστα στα άλλα κράτη. Να σα το παράδειγμα τη Ινδονησία που ήδη αναφέρθηκε. Η Ινδονησία έχει καταβάλει πολλέ προσπάθειε, έχει επενδύσει ιδιαίτερω για να εξυγχρονίσει το, το σύστημα των ενέργειων μεταφορών τη και ω προ το συντονισμό και ω προ την οργάνωση τη ε, υπηρεσία πολιτική αεροπορία και ώστε να ελέγχει καλύτερα τις προδιαγραφές των εκεί εγκατεστημένων αεροπορικών εταιριών. Έχει αποδείξει λοιπόν ότι έχει βελτιώσει σημαντικά σε επίπεδο τεσσάρων της Καρούντα, Airfast, Caron και Premier αεροπορικών εταιριών τις προδιαγραφές με τρόπο που κρίθηκε ικανοποιητικός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τα κρατημέλη και από τον κλάδο της των αερομεταφορών εν γέννη χρειάζονται σημαντικές προσπάθειες και πόροι. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις αρχές και τις αεροπορικές εταιρείε ε, στην Ινδονησία ώστε να ε, διευκολύνουμε περαιτέρω θετικές εξελίξεις. Δηλαδή ενθαρρύνουμε τις χώρες για βελτίωση των προδιαγραφών τους και των συνθήκων ασφαλείας. Η Ινδονησία αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού. Επίσης η ενημέρωση του ε, επιβάτη αποτελεί ιδιαίτερο μέλημά μας τόσο προφορική όσο και γραπτή ενημέρωση κατά τη στιγμή της κράτησης του εισιτηρίου από τον επιβάτη θεωρείται απαραίτητη και θα πρέπει να ενημερώνεται ο επιβάτης από την εταιρεία ότι εφόσον δεχθεί να πετάξει με μια απαγορευμένη εταιρεία παρετείται περαιτέρω δικαιωμάτων του στην συνέχεια. Αλλά επιτρέψτε μου Πρόεδρε να απαντήσω και γραπτό στα λοιπά ερωτήματα γιατί δεν θέλω να καταχρηστώ της ανοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για το θέμα αυτό. Διαδικαστικό, κύριε Σομπερμάγερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άρθρο 173 του κανονισμού. Ένα επεισόδιο που έγινε εδώ πριν από λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στα μονόλεπτα θέματα, Ο κύριος Χαντς Πέτερ Μάρτιν ήρθε και ε, υποτίθεται χιουμοριστικά ε, μας χαιρέτησε με τον χιτλερικό χαιρετισμό. Ε, σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτό αντι, ε, ε, τίθεται και αντίκειται στα ήθη του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ να το ανακαλέσετε στην τάξη και να ελέγξετε εάν μπορεί να τεκμηριωθεί αυτό και από τη μαγνητοφώνηση ή τη μαγνητοσκόπηση. Δεν ξέρω αν αυτοί οι αστεισμοί και οι προκλήσεις έχουν θέσει στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, για την υπόδειξη αυτή. Θα δώσουμε την αντίστοιχη συνέχεια και θα δούμε τι ε, συνέβη. Ευχαριστώ πολύ. So, machen wir weiter in der Tagesordnung. Συνεχίζουμε στη μέση διάταξη. Επόμενο θέμα είναι...